λεπτά για να καταφτάσουμε μεταξύ μας εδώ στην αίθουσα και να υποδεχθούμε την μεγαλειότητα του βασιλεία των κάτω χωρών. Αλεξάνδρ. Ένα λεπτό διάλειμμα.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 μεγαλειότητα είναι μεγάλη μας τιμή που μπορούμε να σας υποδεχθούμε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι άλλωστε παράδοση και σίγουρα μια εξαιρετική τιμή για μας κατά τη διάρκεια της Προεδρίας. Ε, ο αρχηγός κράτους που κατέχει τα ενία της Προεδρίας να απευθύνεται προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε λοιπόν ε, μεγαλειότητα που ε, τηρείτε αυτή την παράδοση. Αποτελείται επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είστε ο πρώτος, το πρώτο, ο πρώτος αρχηγός κράτους ε, της κάτω χωρών που έρχεται να μιλήσει στις, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά είστε ο πρώτος βασιλέας των ε, κάτω χωρών που απευθύνεται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θυμόμαστε την Βασίλισσα Μπέατρεξ, τη μητέρα σας, η οποία μίλησε εδώ στο Κοινοβούλιο και χαιρόμαστε που συνεχίζετε αυτή την παράδοση η Ολλανδική Προεδρία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεργάζονται στενά σε θυελώδεις εποχές. Γι' αυτό χαιρόμαστε λοιπόν και είναι τιμή μας για το γεγονός ότι έρχεστε σήμερα σε τέτοιες θυελώδεις εποχές ακριβώς για να μας απευθύνετε το λόγο. Έχετε το λόγο λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, Ευρωβουλευτές, είναι για μένα ιδιαίτερη εμπειρία να βρίσκομαι ανάμεσά σας κατά τη διάρκεια της Ολλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς είστε οι εκπρόσωποι των πολιτών της Ένωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκπροσωπείτε και αντιπροσωπεύετε τις επιθυμίες τους, τις προσδοκίες τους, αλλά και τις ανησυχίες τους και τους φόβους τους τα ιδανικά τους και τις ελπίδες τους, αλλά και τις ε, απογοητεύσεις τους και το θυμό τους. Όλα αυτά που υποκινούν τους ε, Ευρωπαίους πολίτες ε, ακούγονται και εκφράζονται εδώ. Έχετε ένα σημαντικό καθήκον και ένα δύσκολο καθήκον, ιδιαίτερος τώρα, γιατί είναι πραγματικά άγριος ο άνεμος ο οποίος πνέει στην Ευρώπη. Πολλά από αυτά που για μας ως Ευρωπαίους αξίζουν είναι υποπίεση. Πριν από δύο μήνες αυτή η πόλη, αυτή η γειτονιά επλήχθη από εξτρεμιστικές επιθέσεις στις οποίες έχασαν τη ζωή του 32 άτομα διάφορων εθνικοτήτων και σήμερα σκεφτόμαστε τους ε, συγγενείς τους που έχουν ε, πληχθεί από τον πόνο και τη θλίψη και για αυτούς που εργάστηκαν και εργάζονται για να ανακτηθούν τα όσα χάθηκαν. Οι Βρυξέλλες, η πόλη η οποία είναι στην καρδιά της Ευρώπης επλήχθη, όπως και το Παρίσι πέρσι και τόσες πολλές χώρες κοντά μας και δίπλα μας, η Άγκυρα, το Αχαλέπι, η Βρυτός, η Βαγδάτη, η Σούς, Λαχόρ. Η βία και η καταπίεση καταπιέζουν τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων στην ε, Ευρώπη και γύρω από την Ευρώπη. Και όλες αυτές οι κοινωνίες αποσυντονίζονται. Απελπισμένα πολλοί προσπαθούν και αναγκάζονται να φύγουν και αυτό προκαλεί μεγάλες ε, ροές προσφύγων από το Λίβανο, την Ορδανία, την Τουρκία και πολλές χώρες της Αφρικής και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης νιώθουν και αισθάνονται τις ε, συνέπειες της κρίσης της προσφυγικής κάποιες πιο πολύ από άλλες και η κοινωνική αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών και στο ιστορικό της Ένωσης δοκιμάζονται. Γιατί ο άνθρωπος χρειάζεται μια προστασία, ένα χώρο που μπορεί να αισθανθεί στο σπίτι του. Όπως είπε ο Γερμανός φιλόσοφος Ρίτιγκερ Σαφράνσκι, μπορούμε να είμαστε σε παγκόσμια επικοινωνία και να ταξιδεύουμε παγκόσμια. Δεν μπορούμε όμω να μένουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Μπορούμε να μένουμε μόνο σε ένα συγκεκριμένο μέρο. Και είναι σημαντικό να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι υπάρχει αυτή η συνάφεια, η ανθρώπινη συνάφεια με ένα μέρος. Και για πολλούς Ευρωπαίους η χώρα τους αποτελεί ένα σημείο ε, στο οποίο έχουν ε, ριζώσει. Ένα σημείο, μια χώρα με την ψή της και τα ήθη και τα έθιμά της. Και αυτό ισχύει για τα 17 εκατομμύρια κατοίκους του Βασιλείου της Ολλανδίας, των κατοχωρών. Οι Ολλανδοί ε, αγαπούν τη χώρα τους και είναι περήφανοι για το κλειδοδότημα του, ερασ, του Ερασμού, του Χιούγκο Ντεχρό, του Σπινόσα, του Ρέμπρα, του Φανγκόκ, του Κορνέλης Λέιλε και του Γιώχαν Κράβ. Αλλά με όλη την αγάπη και τη στοργή που έχουμε για τη χώρα μας, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το τι έχουμε και τι οφείλουμε στην γενικότερη ευρωπαϊκή παράδοση και στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, στους λαούς και στους πολιτισμούς γύρω μας γιατί είναι μεγάλες οι αξίε. Οι Έλληνε ήταν εκείνοι οι οποίοι έθεσαν το σπόρο για τη δημοκρατική μορφή του κράτου την οποία διατηρούμε και αγαπούμε. Οι Ιταλοί μα έδωσαν την αναγέννηση, μια πηγή ανανέωση του πολιτισμού και τη επιστήμης. Ο Γάλλο ε, μετανάστη Κριστόφ Πλαντάν ήταν αυτό ο οποίος στο τέλη του 16ου αιώνα δημοσίευσε τα πρώτα λεξικά τη Ολλανδική ε, γλώσσα, Γερμανοί και Γάλλοι φιλόσοφοι όπω ο Λάιπνι, ο Βολτέρο, ε, έθεσαν τι βάσει τη αναγέννηση και του διαφωτισμού. Οι Βρετανοί και οι Πολωνοί σύμμαχοί μα ήταν εκείνοι που μεγάλε θυσίε ε, πολέμησαν για την Ολλανδική ελευθερία το 1944 και το 1945. Τα επιτεύγματα σπάνια, ξέρετε, είναι αμυγό εθνικά. Όσο πιο πολύ ψάχνουμε και όσο πιο βαθιά σκάβουμε, τόσο πιο πολύ υπάρχει σύνδεση των χωρών και των πολιτισμών μα. Και Μπορεί κανείς να περιφράξει μια επικράτεια, όχι όμως ένα πολιτισμό. Η Ευρώπη εκπροσωπεί ένα ιδανικό πολιτισμό προσωπικής ελευθερίας, ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ισότητας και αλληλοκατανόησης. Δύο φορές έχει απευθύνει το λόγο σε σας, στην συνέλευσή σας η μητέρα μου το 1984 και το 2004. Μας υπενθύμησε τις υψηλές προσδοκίες που είχαν στις αρχές της δεκαετίας του 60 πολλοί νέοι σε ό,τι αφορά την Ευρώπη. Αυτό που ξεκίνησε τόσο πεζά όπως ο Χάλιβας και ο Άνθρακας εξελίχθηκε σε ένα κίνημα το οποίο θα καταργούσε τα διαχωριστικά τείχη στην, Ευρώπη, στην Ευρώπη που θα μας εγγυούταν την ειρήνη και θα έδινε νέα δύναμη σε αυτό το τμήμα του κόσμου. Αυτά είχε πει. Εγώ Λοιπόν, γεννήθηκα το 1967. Ένα χαρακτηριστικό και πολύ εντυπωσιακό σημείο στην ιστορία μας και της γενιάς μου ήταν το 1989, όταν τα διαχωριστικά τείχη μεταξύ Ανατολής και Δύσης στην Ευρώπη, τα οποία εμφανόντουσαν πραγματικά αιώνια, ε, έπεσαν. Και το τέλος του ψυχρού πολέμου ήταν η αρχή μιας νέας περίοδου. Και έτσι, λοιπόν... Ε, δημιουργήθηκαν νέοι σύνδεσμοι και έτσι αναπτύχθηκε μία νέα ανατροπία και έτσι άλλαξε η θέση της Ευρώπης στον κόσμο. Μέσα σε μερικές γενιές μόνο η Ευρώπη δεν είναι αυτόματα αυτή που ε, επιτάσσει και προωθεί τη σκέψη. Δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου ούτε από οικονομική ούτε από γεωπολιτική αλλά από πολιτισμική άποψη. Οι αξίε οι οποίε θεωρούμε ότι είναι καθολικέ δεν θεωρούνται αυτονόητε και υπόκειται πιέσει σημαντικέ σε πολλά μέρη του κόσμου. Και ακριβώς όμως επειδή πιστεύουμε στις αξίες αυτές και στην κοινή μας παράδοση, είναι τόσο σημαντική η συνεργασία μας. Γιατί αυτό το επιτάσσει όχι πλέον το παρελθόν, αλλά το μέλλον. Σε τέτοιου καιρού ε, πρέπει λοιπόν να αναρωτιόμαστε τι είδου Ευρώπη ε, αντιπροσωπεύουμε, τι μας κάνει περήφανους. Γιατί συχνά επικεντρωνόμαστε στα προβλήματα, στις ελλείψεις, στις ανησυχίες, αλλά οι ανησυχίες αυτές, έστω και αν είναι δικαιολογημένες και μεγάλες, θα πρέπει να θεωρηθούν στο πλαίσιο των όσων έχουμε πετύχει χάρη στην ευρωπαϊκή συνεργασία. Γιατί ξέρετε, συνηθίζεται εύκολα η ειρήνη. Από τότε που καταρτίστηκε το σχέδιο Σούμαν, κανένα κράτος μέλος δεν έχει στραφεί κατά άλλου κράτους μέλους σε καθεστώς πολέμου, γιατί ε, υπάρχουν πλέον ε, ε, υγιείς σχέσεις εξουσίας. Εγώ είμαι η πρώτη γενιά Ευρωπαίων που συγκαταλέγεται σε αυτή την ευτυχή περίοδο της ιστορίας και το ίδιο εύχομαι και για τις μελλοντικές γενιές. De η επιλογή λοιπόν για την Ευρωπαϊκή Ενωποίηση ήταν μια επιλογή για κοινή κατοχήρωση μιας ελεύθερης και ανοιχτής κοινωνίας με ένα κοινό κρατός δικαίου. 500 εκατομμύρια Ευρωπαίοι καταφέρει να συμφωνήσουν σε μια ένωση κοινών αξιών. Η πραγματοποίηση και η υλοποίηση όλων αυτών γίνεται φυσικά με πολλή συζήτηση και με πολλά συναισθήματα και πολλές, σε πολλές περιπτώσεις εδώ και, και ακόμα και εδώ στο Κοινοβούλιο είναι έντονες αυτές οι διαφωνίες, οι συζητήσεις. Γιατί γίνονται λοιπόν μεγάλες συζητήσεις ό,τι αφορά την μετάφραση αυτών των αφηρημένων αξιών σε συγκεκριμένους νόμους. Και φυσικά είναι μεγάλες και οι διαστάσεις απόψεων. Αυτό σε κάποιες περιπτώσεις θεωρείται αδυναμία της Ευρώπης, αλλά αυτό αποτελεί και απόδειξη της δύναμης της Ευρώπης. Το κριτικό πνεύμα, η ελευθερία ανταλλαγής απόψεων, η συζήτηση, ο δημοκρατικός έλεγχος με κάθε ελευθερία είναι τμήμα της κοινωνίας μας. Μόνο σε δικτατορίες δεν υπάρχει δημόσια συζήτηση. Και γιατί είναι λοιπόν τόσο σημαντικό να συνεχίσουμε μαζί την πορεία μας. Η απάντηση δίνεται κάθε ημέρα από εμάς τους ίδιους. Σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει η έκκληση για καλύτερη συνεργασία και μεγαλύτερη συνεργασία σε ό,τι αφορά τις προσφυγικές ε, ροέ στην καταπολέμηση του ανθρώπινου εμπορίου, τη θερμοκρατία, ε, τη εγκληματικότητα, ε, σε ό,τι αφορά την βελτίωση τη ενεργειακή παροχή, σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση τη αλλαγή του κλίματο, σε ό,τι αφορά τι θέσει εργασία, για 22 εκατομμύρια Ευρωπαίου που είναι άνεργοι και ό,τι αφορά την ενίσχυση τη θέση μα, σε ό,τι αφορά τη καταπολέμηση των δυνάμεων που καταπιέζουν την ελευθερία. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή την συνεργασία. Όπως είπε και πριν από 500 χρόνια ο Έρασμος, τίποτα δεν είναι ευκολότερο από το να νικήσει κανείς τους διαιρεμένους. Η Ευρώπη λοιπόν είναι ενωμένη στην ε, ε, πολυμορφία της και η συνδρομή όλων είναι σημαντική. Το ευρωπαϊκό μπουκέτο λοιπόν δεν είναι ε, πλήρες χωρίς τα ισπανικά λουλούδια, το γαλλικό φλιορδελί, τον άκανθο, τον ελληνικό, την μαργαρίτα της Δανίας, ε, τα γερμανικά ε, και αυστριακά ε, λουλούδια, την κροατική ήριδα, τις τουλίπες της Ολλανδίας και της Ουγγαρίας και το αγγλικό ρόδο ασφαλώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αλλιώς τον κόσμο. Αλλά φυσικά θα πρέπει να υπάρχει κριτική και προς ε, τα όσα συμβαίνουν. Αυτό έγινε και στην ε, κρίση την τραπεζική που αντιμετωπίσαμε και την ανθρωπιστική κρίση μετά από το προσφυγικό, την προσφυγική ροή από την Συρία και άλλες ε, περιοχές. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει γρήγορη αντίδραση από πλευρά τη Ευρώπη. Θα πρέπει να υπάρχει σωστή σχέση μεταξύ τη Ένωση και των κρατών μελών, μεταξύ του Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων, θα πρέπει να συζητάμε τις νέες προκλήσεις και τα προβλήματα. Και παράλληλα υπάρχουν σημαντικές απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τον τρόπο που λειτουργεί η Ευρώπη. Και αυτό ισχύει σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της οικονομίας μας. Η νεολαία μας είναι το μελλοντικό μας κεφάλαιο. Κάνουμε πραγματικά αρκετά πράγματα για να τους δώσουμε επαρκείς δυνατότητες για το μέλλον. Γιατί ό,τι δεν εκμεταλλευόμαστε ως δυναμικό της εσωτερικής μας αγοράς υπολογίζεται σε 1.250 δισεκατομμύρια ευρώ χρόνια μετά την ε, δημιουργία της ενιαίας αγοράς θα πρέπει να μας κάνουν να σκεφτούμε το τι σημαίνει αυτό γιατί η οικονομική και η οικονομική προοπτική για τους καθένα είναι κάτι το πραγματικό και το σημαντικό και αυτό εξετάται σε πολλές περιστάσεις από την οικονομική ανάπτυξη της ε, ενιαίας αγοράς. Η κοινή μας ε, ένωμη αγορά περιλαμβάνει και μια κοινωνική τάξη. Πρόκειται για, τις, για το θέμα των ίσων ευκαιριών, το δικαίωμα να σπουδάσει κανείς, να δουλεύει κανείς, να επιχειρεί κανείς σε ένα άλλο κράτος μέλος, αποτελεί σημαντικό επίτευγμα, αλλά να μην ξεχνάμε και την προοπτική που θα πρέπει να έχουν και αυτοί που μένουν στη χώρα τους, που δεν έχουν ε, τις έξτρα ευκαιρίες, αλλά έξτρα ανταγωνισμό. Γιατί η Ευρώπη για κάποιους σημαίνει το να ανοίγουν τα φτερά τους και για άλλους ε, σημαίνει να υποτάσσονται η ανησυχία πολλών ανθρώπων ίσως σε πολλές περιπτώσεις να συγχέεται με την δυσαρέσκεια με τον τρόπο που, για τον τρόπο που διοικείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούν σε πολλές περιπτώσεις οι άνθρωποι ότι η Βρυξέλλες αποτελεί τον αποτυπωμένο τράγο και ότι ασχολείται με όλα και όχι ότι αποτελεί σύμμαχο. Αλλά όπως στην οικοδόμηση μία ε, καλής γέφυρας θα πρέπει να σκεφτόμαστε τα θέματα ενίσχυσης της βάσης και των θεμελιών λήθων για να μην σπάσει το σημείο αυτό επαφής. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Αυτή η ανάγκη λοιπόν για την ενίσχυση της φέρουσας υποδομής αναγνωρίζεται και στις ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η απάντηση λοιπόν είναι μία. Δεν θέλουμε πιο πολλούς ε, κανόνες, αλλά κανόνες που λειτουργούν καλύτερα επικέντρωση στα βασικά ζητήματα και να λαμβάνονται οι απόψει όσο πιο κοντά γίνεται στον άνθρωπο. Αυτό δεν είναι ενισχύει μόνο την αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά προ... απαντάει και στις ανησυχίες των πολιτών σε ό,τι αφορά την απώλεια της πολιτισμικής τους ταυτότητας. Οι πολίτες μπορούν να θεωρούνται Ευρωπαίοι πολίτες αν αισθάνονται ότι είναι στο σπίτι του στη χώρα του, στην πόλη του στο χωριό του. Γιατί η Ευρώπη ξεκινά, ξέρετε, στο τραπέζι της κουζίνας. Ένας ε, περήφανο Ευρωπαίο είναι και πρέπει να είναι ένα περήφανο Φιλανδό, Γάλλος, Πολωνό, Πορτογάλο, Βρετανό, Βούλγαρος, Έλληνα, Γερμανο ή Ολλανδός. Κανένα, καμία πολιτική τάξη δεν μπορεί να επιβληθεί χωρίς να είναι σε στενή επαφή με το κοινό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι μια ένωση, ένα έργο της ελίτ, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ανήκει σε όλους μας. Ανήκει στον ε, καθηγητή του Πανεπιστημίου, στον οδηγό του λεωφορείου, τον μικρό επιχειρηματία, τον άνεργο, τον ε, συνταξιούχο, τον πρόσφυγα και στα άτομα που δεν έχουν τελειώσει καν το σχολείο. Κάθε χρόνο ένας από τους τρεις, ένας τρεις Ευρωπαίους ε, επισκέπτεται μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Δύο από το πράττουν αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η δική μας, είναι για αυτούς που επιθυμούν να ταξιδέψουν και για αυτούς που μένουν στη χώρα τους. Και έτσι λοιπόν εσείς έχετε μια ιδιαίτερη ευθύνη ως άμεσα αιρετή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώπιον του εκλογικού σας κοινού αλλά και ενώπιον των πολλών που θέλουν να ακουστεί η στην Ευρώπη μέσα των εθνικών ε, εκλογών. Τα αποτελέσματα των ε, ε, εκλογών και των δημοψηφισμάτων και στη δική μου χώρα μπορεί να θεωρούνται πολύ περίπλοκα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά θα πρέπει να μπορούμε να ακούμε το τι λένε οι πολίτες και το εκλογικό κοινό στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Εδώ και 60 χρόνια η ευρωπαϊκή συνεργασία είναι μια γέφυρα που οικοδομούμε προς το μέλλον. Στην αρχή ήταν μικρή η γέφυρα, αλλά με την πορεία των ετών έγινε όλο και πιο ευρία η βάση. Το πακέτο των προδιαγραφών μεγαλύτερο και οι φιλοδοξίες επίσης μεγαλύτερες. Αν θα μπορέσει να μας ε, συνεχίσει να μας υποστηρίζει αυτή η φέρουσα δομή, εξαρτάται από εμά. Όλα εξαρτάται από το κατά πόσο θα κάνουμε, θα είναι αρκετά στενή και ασφαλής και σωστή η σύνδεσμη αυτή. Και είσαστε πάρα πολύ βασικός παράγοντας ως προς την άποψη ε, αυτή ως εκπρόσωποι των πολιτών της Ευρώπης. Αλλά όσο μεγάλη και αν είναι η πολυμορφία και όσο μεγάλες και αν είναι οι διαφορές μας, υπάρχουν πολύ παραπάνω πράγματα τα οποία μας ενώνουν. Σας εύχομαι από βάθος καρδιάς κάθε επιτυχία στο σημαντικό σας καθήκον αυτό.